Procediamo con Επαναλαμβάνεται λοιπόν η συνεδρίαση και να σας ειδοποιήσω ότι με ρητό αίτημα το σύνδεσμο των ε, κοινοβουλευτικών δημοσιογράφων είμαστε υποχρεωμένοι για κάθε αποτέλεσμα ψηφοφορίας να υποδεικνύουμε ρητά τον αριθμό των ψηφισάντων αλλά και των όσων ψήφισαν υπέρ ή κατά. Θέλαμε να απλοποιήσουμε τα... η ζωή μας, αλλά ε, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ψηφίζουμε την έκθεση Κοέλιο για τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχει αποσυρθεί η τροπορφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία, το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 594 ψήφους υπέρ, 51 υπέρ κατά 37 αποχές. Προχωράμε τώρα, συγχαρτήρια καταρχήν στον εισηγητή. Ο κύριος Περόνι παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, διάταξη των εργασιών. Είπατε ότι μετά από αίτημα των δημοσιογράφων, ε, μια καθόλου αξιοσεβαστή κατηγορία, θα ανακοινώνεται όλες τις ψηφοφορίες. Όμως νομίζω ότι ε, ψηφίζουν οι βουλευτές και όχι οι δημοσιογράφοι. Αυτός ο σύνδεσμος των δημοσιογράφων είναι των τυφλών